Um, Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα είναι η συζήτηση για την απαλλαγή 2009 Γενικό Προπολογισμό και μαζί θα κάνουμε κοινή συζήτηση και με όλε τι άλλε απαλλαγέ. Ένα είναι ο συγγητή μα, ο κύριο Όρη. Οπότε, κύριε Όρη, έχετε το λόγο παρακαλώ. Και μετά θα ζητήσω στον κύριο Κατινάλη να πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις απαλλαγές και θα ήθελα να τις συζητήσουμε όλες μαζί ως πακέτο. Έτσι θα εξοικονομήσουμε και χρόνο. Παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Ευτυχώς μπορώ να πω ότι δεν έχω πολλά να πω. Έχω καλά νέα. Δεν έχουμε γενικά σημαντικά προβλήματα. Ούτε εμείς ούτε το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει διαπιστώσει σημαντικά προβλήματα. Ένα γενικό πρόβλημα υπάρχει στο οποίο είχαμε επιστήσει την προσοχή σας και κατά την πρόταση του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λάβουμε τα χρήματα. Όταν έρχεται η ώρα δεν απορροφούνται ε, τα κονδύλια αυτά από τους ε, αρμόδιους φορείς. Δεν υπάρχει δηλαδή απορρόφηση του βαθμού 100%. Τα κονδύλια αυτά στόχο έχουν ε, την προώθηση κοινωνικών θεμάτων και της απασχόλησης. δεν είναι λοιπόν καλό το να μην απορροφούνται η πρώτη μου παρατήρηση. Έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προβλέπετε ότι η απορρόφηση το 2009 ήταν 97,1%. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή απορρόφηση κατά 100%. Έχουν γίνει και λάθη, υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες, ωστόσο πρέπει να διαπιστώσω και αυτό φαίνεται και από την έκθεση, ότι έχουν μειωθεί τα ε, λάθη, το ποσοστό σφάλματος ε, έχει πέσει από 54% το 2007 σε 36%. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η πορεία αυτή είναι θετική. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Ωστόσο, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 βρίσκεται πρώτων θυρών. Ε, υπάρχουν πολλά να γίνουν. Σημαντικό είναι ε, οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιώσουν την ε, απασχόληση. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Έχουμε στόχους όπως είναι η σύγκληση κοινωνική ε, συνοχή κλπ. Μιλάμε πάντα για σημαντικά ποσά εδώ και σημαντικό είναι να θέσουμε τις προτεραιότητές μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προτεραιότητά μας είναι η ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτή είναι θετική τάση. μία έκκληση προς το ελεγκτικό συνέδριο. Να εξετεστούν κονδύλια από τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Με μια σχετική έκθεση θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε γιατί δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως τα κονδύλια. Οι επικρίσεις μου είναι όλες επικοδομητικές. Θα ήθελα να γίνουν ως τέτοιες αντιληπτές. Όσον αφορά ε, τα επιμέρους θεσμικά όργανα, καταρχήν έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, την ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα Ε, επιχειρησιακές δαπάνες ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ χρειάστηκε να ακυρωθούν. Ε, έπρεπε να τηρηθεί η αρχή του ετήσιου χαρακτήρα, θα πρέπει να βελτιωθεί ο προγραμματισμός. Κατά τα άλλα όμως δεν βλέπω να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό ε, αυτού του οργάνου. Μας ε, ενδιαφέρουν οι δραστηριότητες του κέντρου με την Νορβηγία και την Ισλανδία. Πιστεύω ότι η υπηρεσία αυτή γνωρίζει τις απώλειες που έχουν διαπιστωθεί και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διορθωθούν. όσον αφορά το ε, Ίδρυμα του Δουβλίνου. Αρχικά διαπιστώσαμε κάποιες ε, ελλείψεις ε, και κάποιες διαστάσεις απόψεων. Οι ελλείψεις θα πρέπει να διορθωθούν θα πρέπει ε, να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία όσον αφορά το, τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι, ότι οι κανόνες, ότι ο, η δημοσιονομική κατάσταση αποτελεί πολύ ε, ισορροπημένη σειρά κανόνων και δεν ε, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων. Ε, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ε, Ασφάλεια και την ε, Υγεία στην Εργασία. Και εδώ το 18% των πιστώσεων έπρεπε να ε, ακυρωθεί 3,5 εκατομμύρια ευρώ επιχειρησιακών δαπανών έπρεπε να μεταφερθεί στο προσεχές έτος. Ο προγραμματισμός και η εποπτεία είναι το μίσο που υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, ωστόσο έχουμε μια εικόνα που ανταποκρίνεται στην πραγματική δημοσιονομική κατάσταση του οργανισμού αυτού. Οι ε, κανόνες ε, γενικά γίνονται σεβαστοί. Τέλος, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Και εδώ μπορώ να σας πω ότι οι αιτήσιοι λογαριασμοί δεν παρουσιάζουν σημαντικό πρόβλημα, οι κανόνες τηρούνται. Ε, οι συναλλαγές έχει διαπιστωθεί ότι ε, διεξάγονται κανονικά και σύμφωνα με τους κανόνες όσον αφορά την μεταφορά κάποιων κονδυλίων ε, στην επόμενη χρονιά. Αυτό δεν ε, είναι κάτι που επικροτούμε. Σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, Το ελεγκτικό συνέδριο ε, έχει κάνει παρατήρηση σχετικά με την ε, μεταφορά των πιστώσεων. Ο οργανισμός, ωστόσο, έχει λάβει μέτρα ώστε να υπάρχει παρακολούθηση της μεταφοράς, της μεταφοράς αυτής. Πάντως ακολουθείται η σωστή οδός, τηρούνται πιστά οι κανόνες, οι δημοσιονομικοί. Τα, οι διοικητικέ ε, δαπάνες και μισθωτικές δαπάνες είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν, ωστόσο δεν ε, σημειώνονται σημαντικά προβλήματα να συνοψίσω λέγοντας ότι δεν υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Ε, η δημοσιονομική διαχείριση γίνεται κανονικά, δεν έχουμε διαπιστώσει κάποια βασικά προβλήματα. Η γενική μου παρατήρηση είναι ότι δαπανώνται με πολύ λογικό τρόπο, με πολύ φρόνιμο τρόπο η, τα διαθέσιμα κονδύλια. Και σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να διατίθενται. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πεσσινέλη από τον έλεγχο προπολογισμού να μας απαντήσει και στις ερωτήσεις του κυρίου ή να μας κάνετε και ό,τι άλλα σχόλια έχετε παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η Επιτροπή χαίρεται πολύ για τις ε, βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί και που αναφέρονται και στο ελεγκτικό συνέδριο. Η βελτίωση δεν έχει να κάνει μόνο με το ποσοστό σφάλματος, που ίσως είναι ο πιο γνωστός ο δείκτης. Έτσι κι αλλιώς διαφέρει η κατάσταση από χρόνο σε χρόνο. Η βελτίωση έχει να κάνει με όλους τους δείκτες όπως τους αξιολογεί το ελεγκτικό συνέδριο. Για παράδειγμα, ο δείκτης για τους γενικούς διευθυντές που δείχνει τη διαφάνεια και που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά φέτος είναι στην κατηγορία Α, που είναι η καλύτερη κατηγορία. Και όλοι οι δείκτες επίση που είναι στο παράρτημα και δίνει το ελεκτικό συνέδριο δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βρίσκεται σε πολύ καλή υγεία, χέρι πλήρους υγείας. Παρόλο που ανήκει σε μια οικογένεια δύσκολη, γιατί εκεί που έχουμε share management τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν πρέπει λοιπόν να αισθανόμαστε άσχημα, ε, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σφάλμα. Τώρα, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά για τις δυσκολίες ε, χρήσης του προπολογισμού. Οι λόγοι είναι μερικές φορές τεχνικής φύσεως. Για παράδειγμα, το ότι υπάρχει παράτηση της περίοδου εξαιτία της κρίσης της δημοσιονομικής, καθυστέρησαν τα προγράμματα και θα συνεχιστούν το 2011. Όμως ένας από τους λόγους μη πλήρους απορρόφησης είναι και η λιτότητα, μεγαλύτερη λιτότητα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπιστώσει που υπάρχουν λάθη. Και το κάναμε επειδή το ζητήσατε. Το 2008 είχαμε μια δύσκολη στιγμή. Το Κοινοβούλιο για να δώσει την απαλλαγή απίτησε και δικαίω ένα πρόγραμμα δράσης με λιτότητα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έκανε η Κομισιόν λοιπόν. Ακολούθησε και έκανε αυτό που τη ζητήσατε και γι' αυτό είναι σήμερα έτσι η κατάσταση. Πάντως τα πράγματα βελτιώνονται καταλαβαίνουμε ότι φέτος και τις επόμενες χρονιές θα μπορέσουμε να καλύψουμε ε, τις καθυστερήσεις. Αυτά όσον αφορά τα βασικά που είχα να σας πω. Τώρα αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστω είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε. Πρώτα. Α, η κυρία Κόντς πρώτα και μετά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω κι εγώ τη γλώσσα μου. Λέει η κυρία Κόντς. Ως κοιόδης εισηγήτρια θα ήθελα να τονίσω ε, και να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ε, ο Τσάπα Ωρή. Έχουμε εδώ πολύ σημαντικές και καλές προτάσεις από πλευράς του εισηγητή. Θα ήθελα απλά να τις συμπληρώσω σε κάποια σημεία. Ξεκινώ από το από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας. Ο εισηγητής εδώ βασίζεται στις διαπιστώσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις αυτές όσον αφορά ε, το Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Και εδώ ε, συμφωνούμε με αυτά που είπε ο εισηγητής. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο έχει καταβάλει προσπάθειες ε, για να διορθώσει τα, τις ελλείψεις και τα λάθη και να ακολουθήσει σωστή κατεύθυνση. θα υποβληθούν σχετικές τροπολογίες. Όσον αφορά τη... τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ε, συμφωνώ με αυτά που διαπιστώνει ο εισηγητής. Αυτά που έχει πει το ελεγκτικό συνέδριο είναι απόλυτα σωστά. Υπάρχει λόγος όταν κάποιο κέντρο, κάποια υπηρεσία ή κάποιο ίδρυμα δεν μπορεί να απορροφήσει απόλυτα όλους τους πόρους. Ε, αυτό δεν εξαρτάται πάντα από τον ίδιο τον οργανισμό. Θα πρέπει να εξετάσουμε όμως πώς είναι δυνατόν να γίνει καλύτερη χρήση των πόρων. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες ε, εδώ για κάτι τέτοιο. Πάντως ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε και με αυτήν την ε, έκθεση και εδώ θα υποβάλουμε τροπολογία. Γενικά όμως συμφωνούμε με όλες τις θέσεις του εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένη. Δεν άκουσα όλα όσα είχε να πει ο κύριος Όρη, αλλά πώς άκουσα. Συμφωνώ. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι και το είπε ο κύριος ε, Όρη ότι οι συναλλαγές για το γνωσιανοτέτος 2009 σέβονται ε, και τι νομικές πτυχές και είναι όλες τακτικές και νομίζω ότι αυτό αναφέρεται στη γνωμοδότηση. Υπάρχουν ε, κάποια θέματα για τα διάφορα ιδρύματα. Να κάνω ένα-δύο σχόλια και μια-δύο ερωτήσει. Καταρχήν, για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνδικών διαβίωσης και εργασίας. Ε, είδαμε την έκθεση του Λεκτικού Συνεδρίου του 2008 και του 2009 για να δούμε αν διέφεραν τα σχόλια ε, αν το Ίδρυμα είχε υλοποιήσει τις προτάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2008. Εγώ δεν είδα να υπάρχει κάποια παρατυπία εκεί. Κάτι ακόμη σε σχέση με την απάντηση του ίδιου του Ιδρύματος. Ε, λέγεται ότι έχει εφαρμόσει ένα μητρό ξερέσεων από την 1η Ιουλίου 2010, σημείο 15 στην απάντηση. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και θέλω να ρωτήσω πώς κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει εδώ τι σημαίνει αυτό το μητρό εξαιρέσεων και επίσης ε, αναφέρονται και στις διαδικασίες πρόσληψης και στις πληρωμές. Ξέρω ότι και πέρσι υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα με το Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνδικών διαβίωση και εργασία, αλλά ε, διασφάλισαν ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει εφαρμόζοντα τι κατάλληλε δομέ. Έτσι λοιπόν είμαι αρκετά ικανοποιημένη με την απάντηση του Ιδρύματο, αλλά θα ήθελα μία εξήγηση για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσα πριν. Τώρα, δεύτερο σχόλιο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη τη επαγγελματική κατάρτιση, Ευρωπαϊκό Δρόμο Επαγγελματική Κατάρτιση. Πάλι σε απαντήσει του στο Ελεκτρικό Συνέδριο είπαν ότι αποφάσισαν το Μάιο του 2010 επί ενό σχεδίου που θα του επέτρεπε να συμμορφωθούν από το 2013 πλήρω με τι παρατηρήσει του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Και αναρωτιέμαι γιατί θα καθυστερήσουν μέχρι το 2013, πού είναι το πρόβλημα. Και Επίσης χαίρομαι που βλέπω ότι έλαβαν μία απόφαση για να διασφαλίσουν ε, ότι ε, το Συμβούλιο Διαχείρισης θα ενημερώταν για όλες τις μεταβιβάσεις και όχι ε, μόνο για κάποιες που ήταν κάτω ενός συγκεκριμένου κατεφλίου. Αλλά θα ήθελα να λάβω μια απάντηση σε σχέση με την καθυστέρηση αυτή στο το 2013. Και συγγνώμη, ψάχνω τα φαρτιά μου. Ναι, κάτι ακόμα. Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Εδώ δεν έχω ερωτήσεις. Ε, φαίνεται να είναι ικανοποιητικέ οι απαντήσεις. Και για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη τη επαγγελματική κατάρτιση ε, Και πάλι στην απάντηση 13 λέγεται ότι ο σχεδιασμός του προπολογισμού και εκτέλεση του προπολογισμού για το 2009 επλήγει από την αλλαγή της νομικής βάσης του οργανισμού και μετά λέγεται τελευταία στιγμή ε, είχαμε ένα στόλι ενός αποθεματικού 2 εκατομμυρίων. Μήπως κάποιος μπορείτε να μου εξηγήσει γιατί έγινε αυτό και ποιος ήταν ο αντίκτυπος. Περισσότερο θα ακουστώ γιατί βέβαια. Και κάτι Χάρηκα που είδα ότι μας λέει το Ευρωπαϊκό Κέντρο ότι θα ερμηνεύει στενότερα το χρηματοοικονομικό κανονισμό γιατί το Ελληνικό Συνεδρίο ζήτησε κάτι τέτοιο και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Ρή για τις γνωμοδοτήσεις του. Συμφωνώ. Ίσως ε, θα πρέπει να γίνουν μία-δύο τροποποιήσεις, αλλά φυσικά ε, θα τις υποβάλω ανάλογα και με τις απαντήσεις που θα λάβω. Και πάλι ο κύριος Όρη για ενδεχόμενα σχόλια και απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακούστηκαν. ή επίσης μπορείτε να έρθετε και σε συνεννόηση με όποιον έθεσε τα θέματα αυτά. Αυτό εξαρτάται από εσά, ο κύριο Σόρη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Όσον αφορά το Μητρό Εξαιρέσεων, το Register of Exceptions, ειλικρινά δεν γνωρίζω τι είναι αυτό. Δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες όπως η Μαρία, αλλά θα το εξετάσω και θα ε, επικοινωνήσω με τη συνάδελφο. Δεν πιστεύω πάντως ότι αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Η δεύτερη ερώτηση. γιατί το πρόγραμμα αυτό τρέχει μέχρι το 2013. Είναι πολύ δύσκολο το κρίνω εγώ αυτό. Αλλά θα ζητήσω περαιτέρω εξηγήσει και θα μπορέσουμε κατόπιν να αποφασίσουμε πρόβλημα, αν πράγματι μιλάμε για πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα χαρώ πολύ αν οι συνάδελφοι υποβάλλουν τροποποιήσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό θεώρησα το ότι οι οργανισμοί έχουν επικριθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για προβλήματα ελλείψης που υπήρχαν στη δημοσιονομική διαχείριση και έχουν υποσχεθεί να διορθώσουν τα λάθη αυτά. Όλοι όσοι έκαναν τους ελέγχους αυτούς ε, διαπίστωσαν ότι πράγματι η τάση είναι θετική και τα ετρήματα αυτά, τα, οι οργανισμοί αυτοί είναι πολύ σημαντική εταίρια μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πώς τους αντιμετωπίζουμε. Η κυρία Χάρκιν μου έθεσε μια ερώτηση, θα εξετάσουμε αν υπάρχει εδώ πρόβλημα. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ, αλλά θα δώσω πιο συγκεκριμένη απάντηση αργότερα. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Πολύ, Πολύ σύντομα. Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι υπήρχαν και εκπρόσωποι των Ιδρυμάτων όταν συζητούσαμε τα οικονομικά. Νόμιζα ότι θα λαμβάναμε κάποιες εξηγήσει τον Ιανουάριο, λέει πρόεδρο. Α, εντάξει, εντάξει, πολύ ωραία. Ωραία, ευχαριστώ. Ήθελα να σας πω ότι 13 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, υιοθέτηση 1η Φεβρουαρίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Όρη και ας περάσουμε στο επόμενο σημείο για να κλείσουμε και με τη σημερινή ημερησία διάταξη, Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαιδευτική Κατάρτιση για την υποστηρίξη τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Η συγκεκριμένη είναι η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, η έκθεση για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Υποστήριξη της Αττικής Ευρώπη 2020 υπάρχει τώρα. Ε, είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, και η επίσκεψή της στη Σεντεφόπ ήταν πολύ χρήσιμη. Σημαντικό είναι ότι η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να λάβει υψηλή αξία. Πάντα μιλάμε για την εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, αλλά και η επαγγελματική κατάρτιση παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για, στρατηγική Ευρώπη, για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ε, όχι απαραίτητα με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε δηλαδή ανθρώπους με μια ποιοτική εκπαίδευση και ακριβώς ε, γι' αυτό η ποιότητα είναι μια πολύ σημαντική έννοια στην έκθεση αυτή, καθώς ε, και στο σχετικό έγγραφο της Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στην επαγγελματική κατάρτιση. Ε, σημαντικό είναι να λαμβάνει κανείς δεξιότητες σε τέτοιες ώστε να μπορεί αργότερα να μετεκπαιδευτεί. Ε, να λάβει δηλαδή μια βασική εκπαίδευση ε, πάνω στην οποία να βασίσει την περαιτεροπορία του. Σημαντικό είναι αυτό που υπόθηκε και στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, ε, η εικόνα της επαγγελματικής ε, εκπαίδευσης. Σε πολλά κράτη-μέλη η επαγγελματική κατάρτιση θεωρείται κατώτερη. Αποτελεί όμως πολύ καλή εναλλακτική λύση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση εφόσον είναι ποιοτική. Επίσης, μας ενδιαφέρει από την επαγγελματική κατάρτιση να μπορέσει κανείς να περάσει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Για παράδειγμα, κάποιος ε, στη Γερμανία ε, συνηθίζεται όταν έχει ε, επαγγελματική κατάρτιση, όταν έχει γίνει τεχνίτη σε κάποια δουλειά, να μπορεί να περάσει και στο πανεπιστήμιο. Σημαντικό δηλαδή να μπορεί να περάσει κανείς από τον ένα τομέα στον άλλον. Όσον αφορά την ανεργία των νέων, Σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, ε, οι ανθρώπους με ηλικιακή μόρφωση, οι ε, ανθρώπους ε, που δεν έχουν επαρκή κατάρτιση. Υπάρχουν ε, οι απόφοιτοι ηλικίου, οι οποίοι εντάξει κάποια στιγμή βρίσκουν την θέση του στην αγορά εργασία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και με ε, κακή εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Ε, Ενδεχομένω ε, στον επόμενο προπολογισμό να θεσπίσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που να επιτρέπει σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα στι επιχειρήσει, του νέου, στα σχολεία και τι οργανώσει τη νεολαία να δημιουργηθούν δίκτυα που να μπορούν να δώσουν στου νέου αυτού αυτούς κάποια ευκαιρία, διότι ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους αντιπροσωπεύει κάποιο δυναμικό, το οποίο μπορεί να μην αναγνωρίστηκε απαραίτητα στο ε, κανονικό σχολείο. Σημαντικό είναι όταν κοιτάμε τα νούμερα ε, ότι η επαγγελματική κατάρτιση ε, μειώνεται με την ηλικία. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο μέλλον ο κόσμος ε, θα αλλάζει πολύ πιο ε, συχνά εργοδότες ή τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την επαγγελματική κατάρτιση. Προτείνουμε έναν κατάλογο για την επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ελέγξουν τι ζητείτε αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει λάβει καμία μετακπαίδευση και ε, θέλει να ε, κάνει αίτηση για κάποια ε, άλλη θέση εργασίας. Ε, είναι χρήσιμο να γνωρίζει τι θα του ζητηθεί. Ε, είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζει τι επιπλέον χρειάζομαι ώστε να μπορέσω και πάλι να στεριώσω στην αγορά εργασίας. Ε, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει επιγραμμικά, ε, να γνωρίζει κανείς τι χρειάζεται. Χρειάζεται να έχει γνώση υπολογιστών. Ε, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι κάτι πρέπει να κάνω. Δεν αρκεί η πρώτη μου βασική εκπαίδευση. Επόμενο σημαντικό θέμα είναι η ευελιξία και η κινητικότητα. Μπορούμε να επικροτήσουμε ότι, ενισχύονται, ε, ότι ενισχύεται η πρώτη, η βασική εκπαίδευση, ότι ενισχύονται τα στοιχεία αυτά στη βασική εκπαίδευση, ότι πολύ συχνά ήδη από τη βασική εκπαίδευση μπορεί ε, κάποιο ε, σε κάποιο άλλο κράτο μέλο ε, να, κάνει μέρος του, να λάβει μέρο τη επαγγελματική του κατάρτιση ή τη πρακτική του εκπαίδευση. Η στο εξω... παραμονή στο εξωτερικό ε, αυξάνει τις, ε, ε, τις πιθανότητες να το κάνει κανείς αυτό και στο μέλλον. Επίσης υπάρχουν διάφορα μέσα, το Europass, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, τα οποία εξελίσσονται, γίνονται πιο γνωστά και καθιερώνονται περισσότερο. Το Europass, το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο, αποτελεί ε, ιστορία επιτυχίας, όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν αυτό το νέο μέσο. Το άλλο θέμα ε, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο τα κράτη-μέλη είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ώστε να είναι δυνατόν κάποιος σε ένα κράτος μέλος να λάβει την ε, επαγγελματική του εκπαίδευση, σε άλλο κράτος μέλος όμως να πάει να εργαστεί. Ε, εδώ υπάρχει υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να κλείσουν στο μέλλον. Επίσης ε, θα πρέπει να ε, προωθήσουμε ε, το θέμα της τυπικής και άτυπης μάθησης, διότι εδώ υπάρχει τεράστιο δυναμικό το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει αναγνωριστεί. Μία τελευταία παρατήρηση για την χρηματοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σίγουρα αποτελεί εδώ καλό παράδειγμα. Έχουμε όμως εδώ μια ρητή πρόταση τα κάποια κράτη έχουν προχωρήσει στην έκδοση επιταγών κατάρτισης ε, τις οποίες ε, δίνουν σε ανθρώπους ε, με ε, χαμηλό εισόδημα, ώστε να μπορούν ακριβώς αυτές οι ομάδες ανθρώπων να μπορέσουν να μετεκπαιδευτούν. Αυτά πολύ σύντομα. Προσβλέπω στην καλή συζήτηση με τους άλλους βουλευτές και με τους σκιώδεις συζητητές, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα και να δώσουμε την αξία που, στην επαγγελματική εκπαίδευση που της αξίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέντς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δυστυχώς ε, δεν μπορεί ε, να βρίσκεται ο και ο συζητητής του S&D, οπότε θα ε, τον αντικαταστήσω. Ε, χαίρομαι πολύ με την ε, έκθεση αυτή της κυρίας Χίρς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικός τομέας αυτός. Η αύξηση της ανεργίας και οι κοινωνικές συνέπειες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Για να αντιστρέψουμε αυτή την τάση χρειαζόμαστε πιο ευέλικτες μεθόδους και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις νέες συνθήκες ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Φυσικά, το κοινωνικό ταμείο αποτελεί σημαντικό παράγοντα εδώ. Θα υποβάλουμε σχετικές ε, τροπολογίες. Ε, αναφέρθηκε και το European Training Foundation. Ε, εάν δεν κάνω λάθος εδώ στο Κοινοβούλιο, έχει προγραμματιστεί μια διάσκεψη η οποία έχει θέμα την ε, κοινωνική σύγκληση. Βρίσκουμε ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι όλοι στηρίζουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, κύριος ευχαριστώ Ευχαριστώ, κύριε Κυρίε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο την κυρία Χίτς και θέλω να τη συγχαρώ για την εκθεσή της για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό το σχέδιο κειμένου και μπορούμε να δούμε ποιες ε, είναι οι κατευθύνσεις για το μέλλον. Και μπορούμε να δούμε από την έκθεση αυτή ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βάζουμε τη δυνατά μα για να προσαρμόζουμε την επαγγελματική κατάρτιση στι προκλήσει. Ω και όντι εισηγητή, θέλω να κάνω κάποιε προτάσει. Θέλω να ζητήσω από την εισηγήτρια να συμπεριλάβει τα σχόλια μου στην έκθεση πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο των εταιρικών σχέσεων ε, μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, και των επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εταιρικέ σχέσεις ε, όταν μιλάμε για την προσαρμογή αυτής της επαγγελματικής κατάρτισης και επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε στην επαγγελματική κατάρτιση που να αναπτύσσει το επιχειρηματικό πνεύμα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, τους πολίτες ε, να συμμετέχουν σε προγράμματα διαβίου μάθησης. Έτσι λοιπόν ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τέτοια στοιχεία στην έκθεση και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και μία, έκθεση, μία μέθοδο αξιολόγησης αυτής της κατάρτισης. θεωρώ ότι έχουμε καταστήσει και πιο, και πρέπει να καταστήσουμε και πιο ευέλικτη τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, γιατί συνεχώς αλλάζει η αγορά και συνεχώς ε, πρέπει να βρίσκουμε καινούργιους τρόπους χρηματοδότησης της κατάρτισης. Θεωρώ ότι τα σχολεία μου θα εμπλουτίσουν την έκθεση. Είναι πολύ καλή βέβαια η έκθεση και τώρα και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνάδελφος Εμιλή Τουρινέν ε, δεν μπορούσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα και ζητά συγγνώμη. Έτσι λοιπόν ε, παρουσιάζω τα δικά της σχόλια Γενικά είμαστε υπέρ ε, της έκθεσης και πιστεύουμε ότι οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση και θίγει τα περισσότερα κεντρικά ζητήματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία σειρά προτάσεων ε, που, και θεμάτων που θέλουμε να τονίσουμε περαιτέρω. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η επαγγελματική ε, κατάρτιση να είναι δωρεάν και προσβάσιμη σε όλους. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι όταν μπαίνουν στην αγορά εργασίας και την αναγκαιότητα να ε, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους νέους αυτούς στα πλαίσια της επαγγελματική κατάρτισης. Πρέπει να κάνουμε και ένα σύνδεσμο πολύ σημαντικό με την στρατηγική Ευρώπη 2020. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαιδεύση και κατάρτιση» για την υποστήριξη της στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020 και θα θέλαμε δύο ακόμη πράγματα στην έκθεση αυτή. Καταρχήν, πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην επαγγελματική κατάρτιση, αυτό για τους μισθωτούς. Δεν μιλάμε εδώ μόνο για το άτομο, το οποίο πρέπει να είναι υπεύθυνο για την επαγγελματική του εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό αποτελεί κοινή ευθύνη και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν προφανές ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση, γιατί ε, είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των υπαλλήλων τους κάτι που τις αφορά. Και μιλάμε και για τη διαβίου μάθηση. Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει επίσης να αναπτυχθούν σε στενή συνεργασία ε, όλων των ενδιαφερόμενων μέρων, ε, κυρίως ε, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των συνδικάτων και των εργοδοτών. Η αναγνώριση των τυπικών και άτυπων προσόντων είναι θεμελιώδες ζήτημα έχουμε κατά νου να παρουσιάσουμε μία τροπολογία για να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τις καλέ ε, ε, καλές με το μεικτό σύστημα που έχουμε στη Γερμανία και στην Αυστρία και στη Δανία και θέλουμε να καλέσουμε του ε, τους πολίτες να λαμβάνουν υπόψη αυτή την εμπειρία, ε, συγγνώμη, να, να καλέσουμε τα κράτη να λάβουν υπόψη αυτή την εμπειρία κατά τη μελλοντική μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα πρέπει να απευθύνουμε κλεισί σε, στην ε, μάθηση και πρέπει να έχουμε και επαρκή νομοθεσία και ρύθμιση για τη μάθηση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Είναι μια πολύ καλή έκθεση αλλά έχω να κάνω μερικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι που μιλάει για τις δεξιοτεχνίες που απαιτούνται και πρέπει να αναγνωρίζονται ευρύτερα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και η επίσημη κατάρτιση αλλά και η άτυπη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, χαίρομαι που βλέπω στην παράγραφη 24 που αναφέρεται στην διαδικασία της Κοπεχάγης. Είναι ζωτική σημασίας γιατί εφαρμόζεται στην Ευρώπη και γιατί δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη. Αναφέρονται εδώ διάφορα μέσα και τα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μιλάει επίσης για την επαγγελματική κατάρτιση online. Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη, αλλά... Συγγνώμη για το κινητό μου που χτύπησε, λέει η ομιλήτρια. Αλλά είναι πολύ καλό να μιλάμε για τη διαβίου μάθηση και να υπάρχει διαβίου κατάρτιση. Μιλάει επίσης για ένα σύστημα voucher που πιστεύω ότι επίσης είναι θετικό. Πρέπει να δούμε βέβαια τις λεπτομέρειες πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εξαίρετη έκθεση με δύο λόγια και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Δηγάντε, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το έγγραφο αυτό που ετοιμάζεται ε, εκπονήθηκε μετά από την φετινή μας ανακοίνωση. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ σημαντικό για μας, διότι η αρμόδιοι υπουργοί, αρμόδιοι για επαγγελματική κατάρτιση, θα συνεδριάσουν στην Μπρουζ, ακριβώς για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για το σχέδιο έκθεσή σας. Η αξιολόγηση που γίνεται εκεί ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη δικιά μας την ε, αναθεώρηση, η οποία συνδυάζεται με την ε, μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, εν ώψη δηλαδή στρατηγικής 2020, για να είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Η έκθεσή σας υπογραμμίζει τα κέρια ζητήματα. Όντω χρειάζεται να υπάρχουν ευκαιρίε για επαγγελματική κατάρτιση, χρειάζεται ποιότητα, γιατί βλέπετε πολλά από τα πράγματα τα οποία συζητάμε όταν μιλάμε για κατάρτιση είναι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ελκυστικότητα, όταν μάλιστα έχουμε τεράστια ανεργία. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους διαπιστώνουμε στην αγορά εργασίας ότι δεν υπάρχουν οι δεξιοτεχνίες που χρειάζονται για να καλυφθούν οι θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξεπεράσουμε. Μερικά επαγγέλματα θεωρούνται λιγότερο ελκυστικά, παρόλο που δεν έχουν πάντα χαμηλούς μισθούς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τα επόμενα χρόνια αυτό να κάνουμε, να ανυψώσουμε την εικόνα ορισμένων επαγγελμάτων. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να στα επαγγελματικά, μάλλον στις ε, επαγγελματικές δεξιοτεχνίες όταν πρόκειται για κατάρτιση πιο επαγγελματική και λιγότερο θεωρητική πρέπει να ενισώσουμε την εικόνα της. Έπειτα σύνδεση και με τους άλλους τομείς της εκπαίδευσης. Πρέπει να έρθουν οι φραγμοί που υπάρχουν ανάμεσα στην επαγγελματική κατάρτιση και την υπόλοιπη κατάρτιση και μόρφωση. Και να φροντίσουμε, όπως είπα και πριν, να υπάρχουν δεξιοτεχνίες που χρειάζονται. Τώρα δύο σχόλια πάνω στην πρότασή σας. Συμφωνούμε με την έκκλησή σας για να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Σήμερα μάλιστα θα ήθελα να σας δώσω κάποια νούμερα. Καλύπτουμε τώρα για την διασυνοριακή μετακίνηση καλύπτουμε ένα 5%. Με το πρόγραμμα DaVinci που διαχειρίζεται η Επιτροπή, καλύπτουμε ένα 2%. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ μακριά από τον στόχο που είναι 20% των ατόμων στην ανώτατη εκπαίδευση που να μετακινούνται μέσα στην Ευρώπη. Εμεί θα θέλαμε όλοι οι διδάσκοντες στην ανώτατη εκπαίδευση να έχουν αυτή την ευκαιρία να πάνε και να διδάξουν κάπου αλλού. Και οι φοιτητέ πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα βέβαια και να μπορούν όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με φραγμούς και δυσκολίες. Η Επιτροπή στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα προτείνει κάποια benchmarks για την κινητικότητα όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας στηρίξει σε αυτό. Μια δεύτερη παρατήρηση τώρα για αυτά τα βάλουσα τα οποία αναφέρει η συγγήτρια. Η τελευταία πληροφορία που θέλω να σας δώσω είναι ότι σε εποχή κρίσης οι επιχειρήσεις μειώνουν τα κονδύλια που προβλέπονται για την κατάρτιση. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό βέβαια για τις αγορές μας. Η κατάρτιση δηλαδή περιορίζεται στις επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Και δεν θα βγούμε αλλιώ από την κρίση, διότι μειώνοντας τις επενδύσεις στην βελτίωση των δεξιοτεχνών του εργατικού μας δυναμικού δεν θα προχωρήσουμε. Αντίθετα. Αυτή είναι μια πολύ ε, βραχυπρόθεσμη λύση, η οποία όμως δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Ρόλος λοιπόν του κοινωνικού ταμείου πρέπει να είναι τώρα να επικεντρωθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των οικονομιών μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο, μάλλον ερώτηση. Δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι εννοεί η εισηγήτρια στην πρόταση 11 για ένα κατάλογο checklist που λέει όσον αφορά τη διαβίου μάθηση. Τι θέλει να ετοιμάσει η Επιτροπή κάτι τέτοιο για όλες τις χώρες, για όλες τις καταστάσεις και να καλύπτονται εργαζόμενοι που είναι στην αρχή ή στο τέλος του επαγγελματικού τους βίου. Είναι δύσκολο να έχουμε ένα τέτοιο κατάλογο κριτηρίων για τη διαβίου που ζητάει η συγκήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Νάντια Χάρση τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τις προτάσεις. Πολλά από αυτά, πολλές από αυτές μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε. Θα χαρώ πολύ ε, αν ε, λάβω γραπτές ε, τροπολογίες. Ε, δεν είχαμε πολύ χρόνο, γι' αυτό είναι ίσως έτσι τόσο σύντομη η έκθεση. Πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτήν την checklist που αναφέρθηκε, σε αυτόν τον κατάλογο. Υπάρχει, για παράδειγμα, το ευρωδιαβατήριο, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει σε όλες τις γλώσσες. Ε, μπορεί να το βρει κανείς ε, στο διαδίκτυο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς για να παρουσιάσει την ε, σταδιοδρομία του, το βιογραφικό του και την εκπαίδευση που έχει λάβει. Όσον αφορά την μετεκπαίδευση, θα θέλαμε και εδώ να μπορούμε επιγραμμικά να κάνουμε το ίδιο, το ε, πρόσωπο λαμβάνει διάφορε ερωτήσει. Για παράδειγμα, είχατε μετά τη βασική σα εκπαίδευση οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση, ναι ή όχι. Ε, τότε μπορεί να ενημερωθεί κανείς ότι ε, θα, ε, χρειαστεί, θα χρειαστείτε κάποια μεταεκπαίδευση για να προχωρήσετε. Αν κάποιος απαντήσει ναι, τότε ε, ρωτάμε ωραία και πού ακριβώς ήταν η μετεκπαίδευσή σας. Ε, για παράδειγμα, αν ε, κάποιος ε, είναι νοσοκόμος, χρειάζεται άλλη μετεκπαίδευση από ότι κάποιο που ασχολείται με υπολογιστές. Μπορεί λοιπόν να δει κανεί τι δυνατότητες υπάρχουν για μετεκπαίδευση, ποιες δυνατότητες για μετεκπαίδευση έχει ήδη εξαντλήσει ο ετών και έτσι μπορεί να δει ένα χάσμα με προσφορές ε, μετακπαίδευσης ε, τις οποίες ε, να μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θέλει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να υπάρξει μια προσωπική συμβουλευτική συνάντηση στο Γραφείο Ανεργίας ή κάπου αλλού. Νομίζω όμως ότι πρώτο βήμα ε, για τους ε, εργαζομένους ε, είναι να γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται με τις δεξιότητες που έχει, τι μπορώ να κάνω, πού μπορώ να δραστηριοποιηθώ, υπάρχουν άλλες δυνατότητες μετεκπαίδευσης. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Thank you very much for Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 14 Δεκεμβρίου και στις 24-25 Ιανουαρίου θα εξεταστεί από τα μέλη συζήτηση για τις τροπολογίες 15 Μαρτίου υιοθέτηση στην Επιτροπή Πολιτισμού 15 Μαρτίου και υιοθέτηση 16 Μαρτίου. Στις 24 Ιανουαρίου στις 3 θα είναι η επόμενη συνάντησή μας. Ελπίζω όλοι να μπορέσετε να επιστρέψετε. Σας ευχαριστώ και γεια σας.